μερής έρευνα για την εκτέλεση αυτή. Χθε επίσης είχαμε τον πρώτο γύρο πολιτικών εκλογών στην ε, Ουκρανία. Συνάδελφοί μας ε, ήταν παρατηρητές ε, επιτόπου. Δεν έχουμε ακόμα επίσημες πληροφορίες όσον αφορά την διεξαγωγή των εκλογών. Οι συνάδελφοι δεν έδωσαν επισήμως πληροφορίες, αλλά Πρόσεχος βεβαίω θα καταφτάσουν και ελπίζουμε να μας πούν πώ ήταν δίκες οι εκλογές και να γίνει το ίδιο με τον δεύτερο γύρο αρχές Φεβρουαρίου. Από πρώτης πρώτου επίσης η Ισπανία ανέλαβε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ελπίζουμε και με τη νέα συνθήκη να είναι επιτυχής αυτή η Προεδρία και να επιτύχει τους στόχους της. Έχουμε επίσης προγραμματίσει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Ζαπατέρο, ο οποίος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Τρόικας, καθώς δεν είναι μόνο Προεδρία της Ισπανίας, αλλά και του Βελγίου και της Ουγγαρίας. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα να σας ευχηθώ ευτυχές το 2010. Η αρχή της ε, νέας δεκαετίας θα είναι δύσκολη, πρέπει να εργαστούμε σκληρά, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα στις Φρυξέλλες. Έχουμε νέο έτος, νέα συνθήκη, νέα εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει ιδιαίτερη ευθύνη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συνειδητοποιούμε αυτό. Θα ήθελα τώρα να περάσω στην ημερήσια διάταξη. Τα πρακτικά της ε, συνεδρίασης της 17ης ε, Δεκεμβρίου είναι στην διάθεσή σας. Έχετε κάποια παρατήρηση? Αν όχι, εγκρίνονται. Να σας ενημερώσω πως ε, από